Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίσω την έναξη της συνεδρίασης. Όπως γνωρίζετε, την προηγούμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέλεξε το νέο Προεδρείο για την επόμενα δυόμιση χρόνια. Εξελέγει ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι και τώρα ξέρετε ότι με την εκλογή του συναδέλφου Αντώνη Ταγιάννη, το κοινοβούλιο πλέον θα μιλάει πιο πολύ Ιταλικά. Θέλω να συγχαρώ τον ε, κύριο Ταγιάννη για την εκλογή του. Εγώ δεν θα είμαι πρόεδρος, υποψήφιος για πρόεδρος της ε, Επιτροπής ΕΝΒΗ στο δεύτερο ημίση της Διετίας. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές, ε, τη γραμματεία, τις πολιτικές ομάδες του βοηθούς, ιδίως τους βοηθούς μου, την Κάρμεν και τον Ντάριο, για πάρα πολύ επικοδομητική συνεργασία στο πρώτο ήμιση. Ήταν πολύ μεγάλη το προνόμιο και τιμή να προεδρεύω της επιτροπές. Θα συνεχίσω να είμαι τακτικό μέλος και να εργάζομαι με απόλυτη αφοσίωση. Ευχαριστώ πολύ όλες και όλους. Thank excuse me, uh, Chair. Excuse me. Excuse me, Chair, before you... Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, πριν προχωρήσετε δεν γνωρίζω αν αυτό θα είναι ε, το φιλί του θανάτου, θα το πει ένας πράσινος πάντως αυτό, θα το πω. Θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά για τον τρόπο που προεδρεύσατε τα δυόμιση αυτά χρόνια. Ήσασταν δίκαιος, ανοιχτός ε, με τις όλες τις πολιτικές ομάδες και έχετε δημιουργήσει μια πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα στην Επιτροπή μα κάτι που δεν ισχύει σε όλες τις κατανάγκες επιτροπές. Πάντω, σε αυτή την Επιτροπή συνεργαστήκαμε πολύ καλά. Και αυτό παρά τις διαφορές απόψεων μεταξύ μα. Πραγματικά ήσασταν ειλικρινή, τίμιο, δίκαιο πρόεδρος. Ήταν ζωτικό αυτό για την Επιτροπή μα εκ μέρου όλων των συναδέλφων και εκ μέρου των πρασίνων. Και αυτό είναι το φιλθανάτου. Θα μα λείψετε αλλά μην το αναμεταδώσετε αυτό στην Ιταλία γιατί μπορεί να χάσετε ψήφου. Τέλο πάντων, εμεί πάντω σα είμαστε ευγνώμονε. Ευχαριστούμε. Σα ευχαριστώ για τα πράσινα λόγια σα. Λέει ο πρόεδρο. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα ήθελα τώρα να ξεκινήσουμε μια συζήτηση. Οπότε θα περάσουμε στη συνεδρία συγκρότηση σε σώμα, κάτι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας. Να σας υπενθυμίσω ότι ο στόχος είναι να εκλέξουμε τον πρόεδρο και έως τέσσερις αντιπροέδρους ε, για το Προεδρείο της Επιτροπής μας ε, με βάση το άρθρο 24 κανονισμού. Πρώτα εκλέγει το πρόεδρος και εν συνεχεία με τέσσερις γύρους ή τέσσερις αντιπρόεδροι. Έχω ήδη λάβει υπόψη μου τις υποψηφιότητες. Ο κύριο Ζάνη για αντικατάσταση του κύριου Μπρένα. Κυρία Γιάλα είναι σέντερ. Για την κυρία Καμπεθόνα. ο κύριος Φέντρελε, αντί του κύριου Γκερμπράντη. Βόλκεν, αντί Πότς. Πέτερ, αντί Τόλιτς. Γκαρθία Γιλέρα, Αντιβίλμοντ και Ντεμόντε Τζόφι. Και Τζιπ που αντικαθίσταται από την κυρία Ράνθ Γκαρθία. Και ο κύριος Όσλιν, κυρία Όκεν. και Μπαρτ Στάις αντί βαζί. Τώρα λοιπόν μπορούμε να περάσουμε στις ψηφοφορίες δύο. Να σας πενθυμίσω μάλλον ότι για την εκλογή του Προεδρείου. Δεν ψηφίζουμε δυνατά στις χειρός. Όπως δεν έχει λοιπόν την κάρτα ψηφοφορίας, παρακαλώ να λάβει τα μέτρα του ή ώστε κάποιο να του φέρει την κάρτα το συντομότερο δυνατό στην αίθουσα. Γιατί θα είναι μυστική ψηφοφορία. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε αλλιώ. Έχουμε απαρτία. Είναι πάνω από 18 οι παρόντες. Υποψηφιότητες λοιπόν για την θέση του Πρόεδρου. Πολιτικές ομάδες μπορούν είτε και με μονομένοι βουλευτές. Κύριε Λίζε. Ευχαριστώ Τζοβάνι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αλλά στο όνομα του ΕΛΚ θα ήθελα να επαναλάβω αυτό το φίλι του θανάτου από πλευρά των Πρασίνων ε, και νομίζω ε, μιλώ εκ μέρου ε, όλων των μελών τη ΕΝΒΗ. Ήμασταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι με την δουλειά σου ω πρόεδρο. Έχει διευθύνει πολύ καλά την Επιτροπή μας και αγωνίστηκες επιτυχώς για την Επιτροπή μας σε περιπτώσει όπου άλλες επιτροπές ήθελαν να επέμβουν στι αρμοδιότητες μας. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία και χαιρόμαστε που θα παραμείνεις πλήρες μέλος της τακτικό μέλος της Επιτροπής μας και μάλιστα μέλος της Επιτροπής μας με επιρροή και μέλος ε, του Κοινοβουλίου με σημαντική επιρροή. Το αποτύπωμα που αφήνει ε, θα είναι σημαντικό. Νομίζω όμως ότι έχουμε μια πολύ καλή υποψήφιο που θα μπορέσει να ε, πληρώσει τη θέση σου. Η Αντίνα Βαλεάν, που μέχρι τώρα ήταν αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου. και συνόδευσε την προσχώρηση της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει εργαστεί στην Επιτροπή μας και με όλη τη νοσταλγία που νιώθουμε που φεύγει ο Τζοβάνι. Έχουμε αυτή τη φορά μια καλή υποψήφιο και σας παρακαλώ να στηρίξετε την Αντίνα Βαλεάν. Ευχαριστώ. Thank you very much, Peter. Ευχαριστώ, Πίτερ. Έχουμε καμία άλλη πρόταση? Όχι. Νομίζω ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε διαβοή ότι η Αντίνα Βαλιάν γίνεται νέα πρόεδρο της Επιτροπής μας. Καλώ την Αντίνα να προσέλθει στο βήμα και να πάρει τη θέση μου. Καλό απόγευμα, συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας. Έχω συνείδηση της ευθύνης που έχω ως νέα πρόεδρος της Επιτροπής αυτής, που μπορεί να είναι και η πιο σημαντική του Κοινοβουλίου, διότι καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων που έχουν μεγάλη σημασία για τους ε, πολίτες μας ε, και τι εκλογικέ μας περιφέρειες. Ε, προσβλέπω στην καλή συνεργασία με όλους σας και θα προσπαθήσω να ε, στηρίξω και την θέση της Επιτροπής μας εντός του Κοινοβουλίου. Τζοβάνι, σε ευχαριστώ πολύ για την δουλειά που έχει κάνει στην Επιτροπή μας και προσβλέπω στην περαιτέρω συνεργασία. Προχωρούμε τώρα στην εκλογή αντιπροέδρων. Ήδη σημειώθηκε ότι έχουμε απαρτία. Καλό λοιπόν να, να υποβάλλετε υποψηφιότητες για πρώτο αντιπρόεδρο. Παρακαλώ. Ο κύριος Έκχαρτ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, καλώς ήρθατε στην ΕΝΒΗ. Ως πράσινη. Είναι μεγάλη μας χαρά να προτείνουμε τον Βενέντικ Τσαβό που ε, ε, προείδευσε επί μισή χρόνια, ε, μάλλον κράτησε ήδη αυτή τη θέση επί μισή χρόνια. Θα ήθελαμε λοιπόν να το προτείνουμε ως πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής ΕΝΒΗ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Ε, αν όχι, σημειώνω ότι ο κύριος Τσαβό πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Ω υποψήφιο. Ε, τον ε, ερωτώ λοιπόν εάν ε, συμφωνεί με, τη, με τον διορισμό του ως αντιπρόεδρο. Μάλιστα, πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πολύ. Είναι ο μόνο υποψήφιο, οπότε προτείνω να επιβεβαιώσουμε τον διορισμό του διαβοή. Κύριε Τζάβερ, σας καλώ να προσέλθετε στο βήμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, προχωρούμε στον δεύτερο αντιπρόεδρο. Τι υποψηφιότητες υπάρχουν. Παρακαλώ, κυρία Αντέλη. Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς σας ε, συγχαίρουμε για την ανάλυση των καθηκόντων σας. Ε, σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας ε, και προσβλέπουμε στη συνέχιση της καλής συνεργασίας και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον απερχόμενο Πρόεδρο. Προσβλέπουμε λοιπόν ε, στην καλή συνεργασία μαζί σας για τα επόμενα δύο μισή χρόνια. Από πλευρά ε, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για δεύτερο αντιπρόεδρο θα θέλαμε να προτείνουμε την Τατσιάνα Ζάρπου που είχε την ε, θέση αυτή κατά το πρώτο μισό της θητείας αυτής. Καλό λοιπόν τους συναδέλφους να στηρίξουν την υποψηφιότητα. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Αν όχι, σημειώνω ότι η υποψήφια ε, πλήρη τι προποθέσει. Ε, δέχεστε τη θέση αυτή. Ε, ναι, κυρία Πρόεδρε, ωραία. Προτείνω λοιπόν ε, διαβοή να επιβεβαιώσουμε την, την εκλογή τη. Σας καλώ να προσέλθετε στο βήμα και συγχαρητήρια. Τρίτος Αντιπρόεδρος. Η κυρία Ρίτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως συντονίστρια του EFDT στην Επιτροπή αυτή και εκ μέρους της πολιτικής ομάδας θα ήθελα να προτείνω τον Πιερ Νικόλα Πεντιτσίνη ως τρίτο αντιπρόεδρο. Ο Πιερ Νικόλα κατήχε την θέση αυτή τα τελευταία δυόμιση χρόνια και ενημερώθηκα ότι ο Γενικός Γραμματέας ήδη έχει ενημερώσει σχετικά με την υποψηφιότητα αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Υπάρχει άλλη υποψηφιότητα, κυρία Νταλή. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες θα θέλω να προτείνουν τον Πάβελ Πότς για τη θέση του τρίτου αντιπροέδρου. Κατήχε τη θέση αυτή τα τελευταία δυόμιση χρόνια και είναι πολύ δραστήριο μέλος της Επιτροπής αυτής. Θα παρακαλούσα τους συναδέλφους να στηρίξουν την υποψηφιότητα του Πάβελ. Ασθενή σήμερα, δεν είναι παρόν. Έχει ήδη όμως ε, αποστείλει γραπτός ε, τη συγκατάθεσή του για, τον, ε, για την ανάληψη της θέσης. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Όχι, από ό,τι κατάλαβα. Και οι δύο υποψήφοι πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουμε και την συγκατάθεσή τους. Επειδή έχουμε δύο υποψήφιους, θα πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Έχετε όλοι τις ε, κάρτες μαζί σας. Ναι, ωραία. Να πάρω και εγώ τη δική μου. do like this. Um, attribute a color to each candidate. Ε, σε κάθε υποψήφιο θα δώσουμε ένα χρόνο, ένα χρώμα. Θα πρέπει λοιπόν να πατήσετε το ε, κουμπί αυτού του χρώματος. Για τον κύριο Πεντησίνη πράσινο και για τον κύριο Πόρς κόκκινο. Θα πρέπει λοιπόν να πατήσετε πράσινο για τον κύριο Πεντιτσίνη ή το κόκκινο για τον κύριο Πότ. Ανάλογα με την προτίμησή σας. Μία φορά μπορείτε να ψηφίσετε. Εάν θέλετε να απόσχετε, θα τοποθετήσετε την κάρτα στο μηχάνημα χωρίς να ψηφίσετε. Αρχή της ψηφοφορίας. Apparently there is a problem φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μήπως να ελέγξουμε πρώτα, να κάνουμε πρώτα μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Όχι. Ωραία. Είναι ακόμα ανοιχτή η ψηφοφορία. Α, συγγνώμη, πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Δεν φταίω εγώ, συγγνώμη. Παρακαλώ, ψηφίστε πάλι. Αρχίζει πάλι η ψηφοφορία. Δεν ήταν μυστική ψηφοφορία, φαίνεται. Αυτό να ήταν το πρόβλημα. λήξη της ψηφοφορίας. Πενήντα ψήφισαν. Μπορεί να φανεί αυτό στην οθόνη. Βλέπετε το αποτέλεσμα. Με 40 ψήφους εκλέγεται ο κύριος Πότς ως τρίτος αντιπρόεδρος. Θα θέλαμε τον καλέσουμε στο βήμα, δεν είναι παρόν όμως, την επόμενη φορά ίσως. Συγχαρητήρια πάντως. Τώρα έχουμε την εκλογή του τέταρτου αντιπροέδρου. Η κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και πάλι. Εκ μέρου ε, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα ήθελα να προτείνω ως τέταρτο αντιπρόεδρο τον Ζιλ Παρνιό ο οποίος κατήχε τη θέση αυτή τα τελευταία δυόμιση χρόνια. Είναι πολύ δραστήριο μέλος ε, του Κοινοβουλίου και ένα από τα βασικά στελέχη του SND που συμβάλλει στην Επιτροπή μας, ιδιαίτερα σε θέματα που έχουν να κάνουν με την αλλαγή του κλίματος. Θα ήθελα και πάλι να παρακαλέσω τους συναδέρφους να τον υποστηρίξουν. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Νταλή. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Εάν όχι, σημειώνω ότι ο υποψήφιος πληρεί τις προϋποθέσεις. Δέχεται την υποψηφιότητα. Ναι. Έχουμε μόνο ένα υποψήφιο. Προτείνω λοιπόν εκλογή διαβολής. Εφόσον συμφωνείτε. Συγχαρητήρια κύριε Πανιό. Αν θέλετε λάθος το βήμα παρακαλώ.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 σας ευχαριστώ όλες και όλους. Ε, συγκροτήθηκε λοιπόν σε σώμα η Επιτροπή μας. Οπότε μπορούμε να περάσουμε στην ε, κανονική μας ημερήσια διάταξη. Έχω καταρχάς ορισμένες ανακοινώσεις. So, a new point on the approval of the coordinator's recommendation of 12th of January is added as new item. Έχουμε το 7α νέο σημείο, έκριση των συστάσεων των συντονιστών της 12 η Ιανουαρίου. Τώρα αύριο, μετά για τις ψηφοφορίε. αν μείνει χρόνος, παρακαλώ, οι βοηθοί, οι συνεργάτες, λίγη ησυχία παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για αύριο, ώρα της ψηφοφορίας. Εάν μείνει χρόνος, θα έλεγα να συνεχίσουμε μετά την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, να συνεχίσουμε την ψηφοφορία και ίσως και να συζητήσουμε το σημείο 17, ίσως και το 18, μετά το 13, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Εγκρίνεται η για διάταξη με αυτές τις τροποποιήσεις. Ο κύριος Γερμπράντη, τώρα, εισηγητής για τον επιμερισμό των προσπαθειών Effort Sharing, σημείο 10 έχει μπλοκαριστεί λόγω κυκλοφοριακών προβλημάτων και δεν θα έρθει μάλλον το μεσημέρι. Θα έλεγα λοιπόν το θέμα του να αναβληθεί και να μπει στην αυριανή μερισιά διάταξη ως τελευταίο σημείο. Αν συμφωνείτε με την τροποποίηση αυτή. Με αυτές λοιπόν τις τροποποίησεις εγκρίνεται η μερισιά διάταξη. Ευχαριστώ την κυρία Τενμάκη. Τώρα, η αναφορά της αποστολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συνέλευση της ΔΟΠΑ, του ΑΙΚΑΟ δηλαδή, στο Μόντρελ 5 με 7 Οκτωβρίου, έχετε τα έγγραφα στο φάκελό σα, δηλαδή την έκθεση της αποστολής. Η Γενική Συνέλευση λοιπόν του Δεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας εγκρίθηκε στις 6 Οκτωβρίου ψήφισμα για ένα πρόγραμμα μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα για τη διεθνή αεροπορία για την αντιμετώπιση της αύξησης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από την πολιτική αεροπορία στα πάνω από τα 5.020. Επίσης, από τη 1,5-2,5 από τη 1,5 25 απο τη 15 2,5 την, στις 31 Ιανουαρίου έχουμε ένα κοινό εργαστήριο NVITRE για την υποστήριξη της αγοράς για δευτερογενείς πρώτες ύλες οικονομία θα μεταδοθεί ζωντανά. Έχετε επίσης ηλεκτρονικά λάβει τις συστάσεις και αν δεν έχετε παρατηρήσεις θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται επίσης. Σε ό,τι αφορά τι συνεδρία του Οκτωβρίου, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μέχρι τα τέλος, θα θεωρηθούν εγκεκριμένα και αυτά τα πρακτικά. Ολοκληρώνω λοιπόν εδώ τις ανακοινώσεις και περνάμε τώρα στο πρώτο σημείο της μέσας διάταξης που είναι το σημείο 9. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή για του επίσημου ελέγχου 31 Ιανουαρίου και θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ψηφοφορία στην Ολομέλεια έκθεση Κάντενμπαχ. As I said, item 10 will be postponed for tomorrow. Το 10 να βάλετε για αύριο. So we move to item 11 and 12. 11 και 12 μαζί. Τη μελέτη EPRS και το σχέδιο έκθεσης για την οδηγία αποβλήτων σχετικά με τα απόβλητα από ορυχεία. Να ακούσουμε καταρχάς τους εμπειρογνώμονες. Έχουμε τις προσκεκλημένες μας. Θα ακούσουμε την πρώτη. Λοιπόν, Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Πρόεδρε, κυρία Ευρωβουλευτές, ε, το, κλίμα, ε, το τμήμα μας κάνει τις λεγόμενες αξιολογήσεις εφαρμογής με βάση πέντε βασικά κριτήρια, την σκοπιμότητα, συνεκτικότητα, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Όσον αφορά τι εργασίες της Επιτροπής ΕΝΒΗ, ετοιμάσαμε μια τέτοια μελέτη για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα που σας παρουσιάστηκε τον προηγούμενο Μάιο. Η μελέτη για την οδηγία για τα απόβλητα ορυχείων εκπονήθηκε για να υποστηρίξει τις ε, εργασίες σας ε, ε, και είναι ένα θέμα που ορίσκεται στην ημερήσια διάταξη σας σήμερα. Η μελέτη αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο έχει να κάνει με την πρακτική εφαρμογή της οδηγίας με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Το δεύτερο τμήμα εξετάζει τις προοπτικές για την κυκλική οικονομία και θα παρουσιαστεί σε λίγα λεπτά από ε, τον δόκτωρα Έμπερχαρτ Φάλκ και οι δύο παρουσιάσεις ε, θα είναι διαθέσιμες ε, στα ηλεκτρονικά έγγραφα της συνεδρίασης. Να σας παρουσιάσω τα βασικά μας ευρήματα. Καταρχάς να ξεκινήσω από μια σύντομη επισκόπηση της οδηγίας και την εφαρμογή της στα κράτη-μέλη και την υιοθέτηση από διαφόρων μέτρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η οδηγία θεσπίζει μέτρα, διαδικασίες και καθεντήρες γραμμές για να μειώσει στο βαθμό που είναι δυνατόν ε, τα, τις αρνητικές επιπτώσεις ε, από την διαχείριση αποβλήτων ε, από την εξορυκτική βιομηχανία και θεσπίζει απαιτήσει σχετικά με τη διαχείριση των εγκαταστάσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων. Ε, ιδιαίτερα εξετάζουμε τις εγκαταστάσεις κατηγορίας ε, Α, ε, διότι η μη σωστή διαχείρισή τους σημαίνει σημαντικότερους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον. Η προθεσμία για την μεταφορά της οδηγίας ήταν 1η Μαΐου 2008, ωστόσο όλα τα κράτη αντιμετώπισαν προβλήματα και μάλιστα μέχρι το τέλος του προηγούμενου Νοεμβρίου είχαμε και μη συμμόρφωση και μάλιστα τέσσερις εκκρεμείς υποθέσεις ε, με κρατη Έτσι τα περισσότερα κράτη-μέλη ε, δεν έχουν εφαρμόσει όλα σωστά την οδηγία, έτσι δεν υπάρχουν και συνθήκες ίσου ανταγωνισμού. Γι' αυτό η μελέτη συστήνει η εφαρμογή από πλευρά ποιότητα να ολοκληρωθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα για να διασφαλιστούν συνθήκε ίσου ανταγωνισμού για την πρακτική εφαρμογή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, σημαντικά ε, για την πρακτική εφαρμογή είναι κάποια μέτρα που θα πρέπει να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα τα μέτρα της οδηγίας έχουν υιοθετηθεί, εκτός από τις κατευθυντήρες γραμμές ε, για τις επιθεωρήσεις. Και η έλλειψη τέτοιων κατευθυντήρων γραμμών είναι προβληματική, διότι μπορεί να οδηγήσει σε διαφορές όσον αφορά την προσέγγιση στις επιθεωρήσεις από τα διάφορα κράτη-μέλη. Κάτι που φαίνεται και από τα στοιχεία. Έτσι λοιπόν, εάν δεν έχουμε ενιαία εφαρμογή όσον αφορά αυτή την πτυχή, ε, θα δούμε και διαφορά στη συμμόρφωση ε, από πλευρά των οικονομικών φορέων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ω αποτέλεσμα, δεν ε, θα πετύχουν όλα τα κράτη-μέλη εξίσου του στόχου. Με άλλα λόγια, η αποτελεσματικότητα τη πρακτική εφαρμογή θα ποικίλει από ένα κράτο-μέλο σε άλλο. Επιπλέον, η έλλειψη ενιαίων επιθεωρήσεων σημαίνει ότι θα υπάρχουν διαφορέ όσον αφορά το κόστο συμμόρφωση και εφαρμογή. Γι' αυτό η μελέτη συστήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει τις κατευθυντήρες γραμμές για τις επιθεωρήσεις όσο γίνεται πιο σύντομα. Για να έχουμε ενιαία προσέγγιση όσον αφορά τι επιθεωρήσει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να υιοθετήσει τι κατευθυντήριε γραμμέ μέχρι το 2018. Να σα παρουσιάσω τώρα τα βασικά συμπεράσματα όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή τη οδηγία. Τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν έκθεση όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή κάθε τρία χρόνια, συμπληρώνοντα ένα ερωτηματολόγιο. Μέχρι τώρα δύο φορέ ε, έχει γίνει αυτή η έρευνα που καλύπτει την πρακτική εφαρμογή ανάμεσα στο 2008 και το 2014. Αξιολογήθηκε η ποιότητα των ε, δεδομένων που υποβλήθηκαν πέρσι το Σεπτέμβριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η Επιτροπή ΕΝΒΙ συζήτησε με την Επιτροπή πάνω στο θέμα αυτό τον Νοέμβριο. Η ιδιαίτερη Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα ε, δεδομένα δεν αρκούν για να έχουμε μια ε, επαρκώς ε, λεπτομερή και αξιόπιστη εικόνα. Επιπλέον, τα κράτη-μέλη υποβάλλουν εκθέσει σχετικά με τα μέτρα που έχουν υιοθετήσει, όχι όμω σχετικά με την πρακτική του εφαρμογή. Και η μελέτη μα διαπίστωσε ότι το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε επίση έχει κάποιε ελλείψει και έτσι δεν είναι αρκετά καλή η ποιότητα των δεδομένων. Σημαντική έλλειψη που θα πρέπει να αναφερθεί είναι ότι το ερωτηματολόγιο δεν επιτρέπει την εφαρμογή την δημιουργία βάσης δεδομένων ε, σχετικά με τις εγκαταστάσεις ε, στον χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι τα κράτη-μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν ακριβή αριθμό εγκαταστάσεων και να ε, που που ακριβώ βρίσκονται εντό του εδάφου του. Και χωρί μια τέτοια βάση δεδομένων ε, που να καλύπτει το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, η πρακτική εφαρμογή τη οδηγία θα είναι ελλειπή. Και γι' αυτό η μελέτη συστήνει να βελτιωθεί αυτό το σύστημα ερωτηματολογίων ανά τριετία. Ιδιαίτερα δεδομένου ότι η τρίτη αυτή προσπάθεια θα ξεκινήσει τον Μάιο. Ανάμεσα στα 2008 και το 2014 διαπιστώσαμε τα εξής προβλήματα. Καταρχάς, κατηγοριοποίηση των εγκαταστάσεων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Ιδιαίτερα όχι τις εγκαταστάσεις κατηγορίας Α. Εάν δεν γίνει σωστή καταγοριοποίηση μιας εγκατάστασης επεξεργασίας ε, αποβλήτων, σύμφωνα με την οδηγία, αυτό σημαίνει ότι η εγκατάσταση αυτή δεν ε, θα ε, πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις της οδηγίας ή στις πιο ειδικέ ε, προϋποθέσεις εάν θεωρηθεί εγκατάσταση κατηγορίας Α. Και αυτό θα ε, έχει συνέπειες όσον αφορά την ασφάλεια. Το δεύτερο πρόβλημα σχετίζεται με τις άδειε. Κάποιες εγκαταστάσεις είτε λειτουργούν χωρίς άδειε ή δεν συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην άδεια που έχει χορηγηθεί και ιδιαίτερα για ε, καταστάσεις κατηγορίας Α. Το πρόβλημα συνδέεται ε, με την έκδοση αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Τρίτο πρόβλημα είναι οι διάφορες προσεγγίσεις που ακολουθούνται από τα κράτη-μέλη όσον αφορά τις επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων. Δεύτερη προβληματική πτυχή είναι ότι εξωτερικά μέτρα ε, επίγουσας ανάγκης λείπουν για το 25% των εγκαταστάσεων κατηγορίας Α που έχουν ε, υποβληθεί από τα κράτη-μέλη. Τέλος, ε, ανάμεσα στο 2008 και στο 2014 είχαμε πέντε ατυχήματα σε ευρωπαϊκό έδαφος και έξι διαδικασίες επί παραβάση για κακή εφαρμογή. Περισσότερες λεπτομέρειες ε, μπορείτε να διαβάσετε στην μελέτη. Συστήθηκε τα προβλήματα που εντοπίστηκαν να αντιμετωπιστούν από τα κράτη-μέλη επιγόντως. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η μελέτη μπόρεσε να αξιολογήσει την εφαρμογή με βάση μόνο τρία κριτήρια. Τη σκοπιμότητα, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα. Ιδιαίτερα, ενώ η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων ε, ε, ανταποκρίνεται στις ανάγκες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι ε, επικύλουν τα επίπεδα αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή από, την, από τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Φάλκ που θα σας μιλήσει για τις προοπτικές, για τις εξορυκτικές δραστηριότητες στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο. Όπως ξέρετε, ε, ε, έχετε το λόγο τώρα, κύριε Φάλκ, για να μας μιλήσετε για την θέματα κυκλικής οικονομίας σε σχέση με τις ε, εξορρυκτικές βιομηχανίες και τις μονάδες αποβλήτων. Θα σας μιλήσω για αυτή τη μελέτη που προετοιμάσαμε πέρυσι επί του θέματος. Ελπίζω να ανταποκριθώ γιατί έχω ορισμένα προβλήματα με τις διαφάνειες. Θα ήθελα να ε, ξεκινήσω με μια θαραλέα δήλωση, ίσως και προκλητική, γιατί νομίζω ότι όλες οι διαδικασίες εξόριξης είναι ε, σώστες εάν ακολουθήσουν τις ε, καλύτερες πρακτικές και τις συστάσεις περί αυτών. Και αυτό σημαίνει ότι ο ρυθμιστής θα πρέπει να ορίσει πολύ καλύτερα αυτό το πλαίσιο. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο καλά όσο θα έπρεπε, γιατί υπάρχει πίεση από την ε, οικονομία και επειδή υπάρχουν και πολλές ε, παραβλέψεις στα πλαίσια των, της επίβλεψης και επίσης έχουμε να κάνουμε με εγκαταστάσεις για τις οποίες ε, δόθηκε άδεια όταν οι χρηστές πρακτικές ήταν εντελώς διαφορετικές και οι οποίες έχουν πλέον εξεπεραστεί. Επίσης, τα προβλήματα σχετίζονται με το γεγονός ότι γίνεται κατακράτηση μεγάλου, ε, μεγάλου αριθμού αποβλήτων υπό υγρή μορφή και αυτό έχει ε, σημασία ιδιαίτερα για τα φράγματα τα οποία ε, κατακρατούν πολύ νερό. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να λάβουμε υπόψη αυτές τις δεξαμενές συγκράτησης καταλήπων και να ανταποκριθούμε καλύτερα στη διαχείρισή τους. Θα πρέπει λοιπόν να μειωθεί το περιεχόμενο σε ε, είδωρ. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ενέργεια. Άρα θα πρέπει να εξοικονομήσουμε ε, τα πλαίσια δημιουργίας, μάλλον χρήσης ενέργειας και βεβαίως τους ε, κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουμε. Επίσης δεν πρέπει να εξορίσουμε υλικά που δεν είναι απολύτως αναγκαία. Επίσης το, ε, το υλικό αυτό θα πρέπει πολλές φορές να μην φτάσει μέχρι το επίπεδο της γης, δηλαδή να αφήσουμε ε, αυτό το υλικό στις υπόγειες αυτές δεξαμενές. Κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει βεβαίως και προβλήματα τεχνικής φύσης. Ποιες είναι οι εναλλακτικές μέθοδοι που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στην περίπτωση συγκράτησης καταλήπων αυτό που έχει λοιπόν σημασία είναι να κρατήσουμε αυτά τα κατάλοιπα κάτω από τη γη, μέσα στα πλαίσια της χρήσης αυτών των δεξαμενών. Και μπορούμε πολλές φορές in situ επιτόπια να κρατήσουμε αυτά τα υλικά υπογείως. Υπάρχουν και άλλα υλικά ή πρώτες ύλες που μπορούμε να εξορίξουμε μέσα στα πλαίσια μιας διαδικασίας εξόριξης που είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμη. Αυτό μπορούμε να το δούμε μόνο αναπερίπτωση. Επίσης, πολλές φορές θα πρέπει να αλλάξουμε τη διαδικασία, διαδικασία δημιουργίας καταλήπων και αποβλήτων. Θα πρέπει να έχουμε μια συνεκτική διαδικασία εξόριξης, έτσι ώστε να κρατάμε αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι πραγματικά αξιόλογα Δηλαδή φέρνουμε αυτές τις πρώτες ύλες ε, στην ε, ε, επίγεια επιφάνεια και χρησιμοποιούμε τα υλικά τα οποία πραγματικά είναι χρήσιμα. Δηλαδή δεν θα ήταν σκόπιμο ορισμένα βαρέα μέταλλα να φτάσουν στην επιφάνεια της γης, κάτι το οποίο θα μπορούσε να σημαίνει κίνδυνο για το περιβάλλον. Εάν λοιπόν μπορέσουμε να διαχωρίσουμε τον τομέα των αποβλήτων και της εξόριξης καθεαυτής, αυτό θα βοηθούσε την ε, ανάκτηση αργότερα, αν υπάρχουν στοιχεία στα κατάλοιπα τα οποία θα ήταν ενδιαφέροντα, θα παρουσίαζαν ενδιαφέρον. Όμως αυτές οι διαδικασίες χρειάζονται συστημική αποτίμηση σε σχέση με τις ανάγκες ενέργειας για να υπάρχει ευεργέτημα αν αλλάξουμε αυτές τις αλυσίδες εφοδιασμού και επίσης να μην υπάρξει ρήξη σε αυτή την αλυσίδα γιατί υπάρχουν και κρίσιμες ομάδες που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και φυσικά όλα αυτά θα πρέπει να είναι βιώσιμα ε, στα πλαίσια της ε, συνολικής οικονομικής συγκυρίας. Διαφορετικά δεν έχουν νόημα. Φτάνουμε στην κυκλική οικονομία, σε αυτό το πρότυπο, το οποίο μας απασχολεί σήμερα. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι οι θερμοδυναμικές αρχές μας δείχνουν ότι κάθε διαδικασία οδηγεί σε απώλειες. Θα πρέπει λοιπόν να τις περιορίσουμε. Επιπροσθέτως, οποιαδήποτε διαδικασία σημαίνει ότι θα υπάρχει εισρωή ενέργειας και γι' αυτό ε, θα πρέπει να δούμε αυτή την κυκλική διαδικασία η οποία είναι αναπόφευκτη να δούμε ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά, να γίνει σωστή χρήση των ε, ορυκτών ε, πόρων και να μειώσουμε το αποτύπωμα του άνθρακα. Επίσης, ορισμένα σύγχρονα υλικά είναι δύσκολο να ανακυκλωθούν, διότι προαπαιτούν ε, υψηλή χρήση ενέργειας, δηλαδή χρειάζεται πολλή ενέργεια για να διασπάσουμε αυτά τα υλικά. Η ανακύκλωση λοιπόν αφορά και τα κατάλοιπα, τα ορυκτά κατάλοιπα και θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα θετικά στοιχεία. Θα ε, φτάσουμε σε μια βιώσιμη αγορά και θα ε, επιβαλόταν να έχουμε πολύ χαμηλότερο αποτύπωμα διοξίδιου του άνθρακα. Επίσης θα ε, πρέπει να προωθήσουμε την αρχή της ενδυνάμει ε, απομάκρυνσης του κινδύνου ή μεταφοράς του κινδύνου αλλού. Θα πρέπει να υπάρχει ε, ένας συστηματικός και συστημικός κύκλος ζωής, μια αξιολόγησή του, για να δούμε ποιες είναι, ποια είναι η σχέση κόστους ωφελίας. Και μόνο τότε θα πρέπει να προωθήσουμε αυτή την ανακύκλωση και να δώσουμε και φορολογικά κίνητρα. Ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτής της ε, πολιτικής. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η εξόριξη και η διαδικασία ε, επεξεργασίας δεν λαμβάνει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον. Εξαρτόμαστε πλέον από τις εισαγωγές και η εξόριξη γίνεται σε τρίτες χώρες. Όταν δούμε λοιπόν τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τη διαχείριση καταλήπων, θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει αλλού. Φτάνουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις αυτές κινούνται στο εξωτερικό, εκεί που δεν υπάρχει τόσο αυστηρή ε, νομοθεσία και όπου υπάρχουν περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι υγείας, πολύ ψηλότεροι από ό,τι στην Ευρώπη. Επίσης, όταν παρεμβαίνουμε στην ε, δημιουργία μιας πολιτικής και προώθησή της, τότε επεμβαίνουμε, είμαστε παρεμβατικοί ως προς την ε, ελεύθερη οικονομία της αγοράς. Θα πρέπει, συνεπώς, να έχουμε ε, αξιολογήσεις αντικτύπου, οι οποίες να είναι συνεκτικές και συστηματικές εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα για να αποφύγουμε τις αδόκητες συνέπειες. Γιατί πολλές φορές υπάρχουν βραχυχρόνια ευεργετήματα, αλλά όχι μακροχρόνια για την οικονομία και για την ανθρωπότητα γενικότερα. Για να φτάσω σε ε, ορισμένα συμπεράσματα θα ήθελα να πω τα εξής. Πιστεύω ότι η εξόριξη έχει μεγάλη σημασία ε, στην ε, οικονομία μας, για την οικονομία ενός βιομηχανικού κόσμου και ακόμα και όταν θέλουμε να είμαστε πιο αποτελεσματική θα πρέπει να μην υπάρχει, να, μάλλον να περιορίσουμε τη διαδικασία διάχυσης, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε αυτοκίνητα. Υπάρχουν πολλά υλικά τα οποία φτύρονται από τη σκουριά, η οποία στη συνέχεια δεν μπορεί, αυτά τα υλικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανακύκλωση. Υπάρχουν λοιπόν απώλειες τις οποίες θα πρέπει να περιορίσουμε. Επίσης, οφείλουμε να δούμε ποια στρατηγική είναι η πιο αποδοτική και ποια είναι εκείνη η οποία ενέχει χαμηλότερο οικονομικό κόστος και μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Θα πρέπει να ορίσουμε αυτές τις δαπάνες σε σχέση με την όλη διαδικασία διατήρησης και ανακύκλωσης των υλικών. Και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όχι μόνο αποτυπώνουμε, διατυπώνουμε κανονισμούς, αλλά επιβάλλουμε στους ρυθμιστές να εποπτεύουν αυτούς τους κανονισμούς, γιατί με με λιγότερη εξόριξη, σε χώρες όπου υπάρχει λιγότερη εξόριξη, ο, ο ρόλος του ρυθμιστή έχει αποδυναμωθεί και φυσικά δεν υπάρχει και η κατάλληλη τεχνογνωσία πάντα ή μειώνεται. Εάν λοιπόν προωθήσουμε εναλλακτικές ε, διαδικασίες θα πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμες. Διαφορετικά η βιομηχανία δεν μπορεί να επιβιώσει και πάει στο εξωτερικό, μετακινείται στο εξωτερικό με τις συνέπειες που σας προανέφερα. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Σίγουρα στη συζήτηση θα προκύψουν ερωτήματα. Ευχαριστώ και εκ των προτέρων που θα παραμείνετε εδώ για τη διάρκεια της συζήτησης, όπως προείπα. Έχουμε ένα σχέδιο έκθεσης για την εφαρμογή της οδηγίας που θα συζητήσουμε. Ο κύριο Αλβενή, που είναι ο συγγετή μα, θα πάρει πρώτο το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που έφτασα την κατάλληλη στιγμή στην Επιτροπή περιβάλλοντος. Είχαμε μία μακρά προπαρασκευαστική περίοδο και τώρα ήρθε η στιγμή επιτέλους για μία σε βάθος συζήτηση περί της εφαρμογής της οδηγίας για τα πόβλητα ορυχείων. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τη μονάδα Expo Post Impact Assessment ε, από το ΕΠΑΡΕΣ e την κυρία Καραμφίλογα αλλά να ευχαριστήσω και τον κύριο Φάλτο, αν ξέρω τον προγνώμη. Ήταν πάρα πολύ καλή η μελέτη αυτή και σίγουρα θα βοηθήσει και εμάς, γιατί ήταν πραγματικά ένα δύσκολο εγχείρημα εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Πρόσωποι της των πολιτών έχουν επίσης τοποθετηθεί, υπήρξαν διαβουλεύσεις και με άλλους φορεί. και πραγματικά πρέπει να τονίσουμε το ρόλο των οργανισμών των πολιτών που έδωσαν πολύτιμη συνεισφορά για την έκθεση αυτή. Το είπα και στην ανταλλαγή απόψεων που είχαμε το Νοέμβριο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εδώ και πολύ καιρό η εξωτερικές δραστηριότητες προς εκείνο το ενδιαφέρον μας. Έχουμε αντιμετωπίσει διάφορα ζητήματα, έχουμε συζητήσει αναφορές ε, πολιτών, ε, έχουμε θέσει στην Κομισιόν διάφορα ζητήματα. Έχουν γίνει ακροάσεις και διάφορες άλλες συζητήσεις. Όπως επίσης έχουν εγκριθεί και πολλά ψηφίσματα τα τελευταία χρόνια. Και η οδηγία θεωρείται ένας τομέας ιδιαίτερα ενδιαφέρον από πολλές από αυτές τις αναφορές ψηφίσματα κτλ. Και δει η εφαρμογή της οδηγίας και η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο Άλλωστε αυτό είναι και μέσα στο δικό μας πεδίο αρμοδιοτήτων. Είχαμε και τη μελέτη για την εφαρμογή. Μας βοηθά πολύ ε, η μελέτη και εγώ θα σας πω τώρα και τα βασικά συμπεράσματα στη μητρική μου γλώσσα, όμως τα ουγγρικά. Οπότε βάλτε και ακουστικά παρακαλώ. Έχουμε λοιπόν την ε, προθεσμία του 2018 για την εφαρμογή της οδηγίας, αλλά υπήρξαν καθυστερήσεις ε, και έχουν ε, κινηθεί και διαδικασίες επί παραβάση. Οπότε δεν αναμένουμε όλα τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να εφαρμόσουν έγκαιρα αυτή την οδηγία. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε επίσης. σε ό,τι αφορά την πρακτική εφαρμογή του ελέγχου. Και αυτό είναι προβληματικό. Με βάση τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα, φαίνεται ότι τα κράτη-μέλη έχουν να αντιμετωπίσουν πρακτικέ δυσκολίε σε ό,τι αφορά τι αδειοδοτήσει, τον έλεγχο. Εξωτερικό, εξωτερικά σχέδια κτλ. Με τι γενικέ κατευθυντήριε γραμμέ τη Κομισιόν θα βελτιωθεί η κατάσταση και πιστεύω ότι θα διορθωθούν και ορισμένα από τα προβλήματα. Όμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει και άλλα. Έχει δώσει διάφορα ε, έγγραφα στη δημοσιότητα. Ένα από αυτά έχει να κάνει με τις αρμοστικές διατάξεις ε, και υπάρχουν και κατευθυντήριες γραμμές όμως για τους έλεγχους που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Λείπει αυτό το σημαντικό έγγραφο. Και αν δεν υπάρχει ένα απλό, ένα νέο πλαίσιο για τους ελέγχους, θα υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα, γιατί θα βλέπουμε σημαντικές αποκλήσεις ανάλογα με το κράτος μέλος. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συντομότερο δυνατό θα πρέπει να προχωρήσει στην έγκριση των γενικών αυτών κατευθυντήρων γραμμών. Σε ό,τι αφορά τώρα το σύστημα υποβολής εκθέσεων αναφορών, δεν πληρεί το σκοπό μιας συνέχεια μιας παρακολούθησης και αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν ελλείψεις Σε ό,τι αφορά δε το ερωτηματολόγιο ιδίω ε, και θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να διορθωθεί το πρόβλημα. ώστε να ισχύσει το νέο πλαίσιο κατά την ε, εφαρμογή και όχι το παλαιότερο που παρουσιάζει προβλήματα. Υπάρχουν δυσκολίες, ε, υπάρχουν διάφορες εγκαταστάσεις, μονάδες, ε, πρέπει να καταγραφούν. Επειδή υπάρχουν όμως προβλήματα, δεν μπορούν να καταγραφούν και ε, επομένως και να παρακολουθηθούν όλες αυτές οι εγκαταστάσεις, ούτε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις αρνητικές επιπτώσεις των αποβλήτων στις τοπικών κοινωνιών και το τονίζω, τοπικών κοινωνιών έχουμε και τη σχέση κόστος-οφέλους. Μέχρι τώρα δεν είχαμε την απαραίτητη προσοχή σε προληπτικά μέτρα. Ούτε οι τοπικές κοινωνίες, οι τοπικές αρχές συμμετείχαν. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή και σε αυτό το επίπεδο. Διότι τα απόβλητα ορυχείων είναι το 1 τρίτον του συνόλου των αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρόλα αυτά δεν δόθηκε η επαρκής προσοχή ούτε από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επεξεργασία αυτών των αποβλήτων μπορεί να ενταχθεί όμως στην κυκλική οικονομία. Όμως, στο πακέτο του 2015 για την κυκλική οικονομία δεν περιλήφθη αυτό το στοιχείο. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι πρέπει να περιληφθεί να περιληφθούν δηλαδή τα απόβλητα ορυχείων στην κυκλική οικονομία. Αυτό απαιτεί πολιτική απόφαση. Αλλά θα επηρεάσει θετικά και την επεξεργασία των αποβλήτων αυτών, άρα θα έχει θετικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα. Με βάση τη μελέτη, τεχνολογίες που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, είναι όριμες, είναι ασφαλείς. Αλλά μόνο εφόσον βέβαια πληρούνται όλοι οι όροι και όλες οι υποθέσεις Υπάρχει, επαναλαμβάνω, μεταξύ του τι είναι προβλεπόμενο και του τι γίνεται στην πράξη μια μεγάλη απόσταση. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Και πολλές φορές παραγνωρίζονται ορισμένοι κανόνες. Ορισμένες μονάδες για χρόνια και δεκαετίες λειτουργούσαν με βάση πρακτικές που δεν συμβαδίζουν με τις απαιτήσει ε, τις Και φυσικά για τον εξυγχρονισμό των μονάδων αυτών απαιτούνται τεράστιες ε, επενδύσεις. Νομίζω ότι η έννοια της καλύτερης δυνατής ε, τεχνολογίας, ε, η βέλτιση πρακτικής είναι κάτι που θα πρέπει να το ξαναδούμε. Γιατί θα πρέπει να αποφύγουμε την εφαρμογή πρακτικών που δεν είναι αυτής της τελευταίας, αυτές της τελευταίας αιχμής τεχνολογίας, αλλά οι πιο καθιερωμένες ε, ε τεχνολογίες. Ε, υπήρξε ένα ψήφισμα το 2010 για την ε, κατάργηση μιας πρακτικής συγκεκριμένα. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη λοιπόν οι τελευταίες εξελίξεις, ε, τελευταίες μελέτες και να αντλούνται διδάγματα από τις διάφορες φυσικές καταστροφές ή καταστροφές ό,τι αφορά την απόθεση αποβλήτων. Θα πρέπει λοιπόν να ιεραρχήσουν σωστά τι προτεραιότητες, βάζοντα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας σε πρώτο πλάνο, ακόμη και αν μπορεί η σχέση να μην είναι η βέλτιστη δυνατή. Επίσης πρέπει να τηρούνται αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα. και να επιλέγεται η καλύτερη επιλογή για το περιβάλλον παρότι μπορεί να είναι πιο δαπανηρή από άλλες. Δεν έχω πολύ χρόνο για να μπω σε άλλες λεπτομέρειες ό,τι αυτά τα πορίσματα της μελέτης. Όμως, αν μου επιτρέπετε, κλείνοντας, να πω ότι για μένα η πραγματική επίπτωση ε, ατυχημάτων ή καταστροφών ήταν η απόλυτη αποτυχία της αρχής ο πληρώνει. Διότι, ναι μεν, Υπάρχει σχετική ρήτρα στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αν όμω δεν υπάρχουν εχέγγυα και εγγύσει, δεν μπορούν οι ρηπαίνοντε τελικά να καλύψουν το κόστος που προήλθε από την αμέλειά του. Και επομένως, αναπόφευκτα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει το έργο της προς ε, ένα σύστημα εγγύησης ε, προστασίας από ε, βιομηχανικές καταστροφές και ατυχήματα, ώστε να μπορεί ο Ριπένον στην πράξη να πληρώσει σε περίπτωση μιας μεγάλης καταστροφής. Είναι κοντά μας η λύση. Καιρός είναι λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τις ευθύνες της σε αυτό το επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χολγενή. Η κυρία Ντάλη από το S&D. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι παρόντες και μας δίνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Μιλώ εκ μέρους του σκιώδου συζητητή μας, του κυρίου Νίκολα Καπούτο, που δυστυχώς δεν μπόρεσε να παραβρεθεί εδώ σήμερα. Σας παρουσιάζω λοιπόν και τη δική του θέση πάνω στην έκθεση και το θέμα αυτό. Θα θέλαμε καταρχάς να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κολβένη για την εξαιρετική έκθεση, η οποία θίγει όλα τα βασικά σημεία της σχετικής οδηγίας. Το πιο προφανές που αναφέρθηκε είναι η καθυστέρηση και η κακή ποιότητα κατά την μεταφορά της οδηγίας αυτής. Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις η οδηγία ε, ισχύει πάνω από τα δύο χρόνια που προβλέπονταν. Αλλά γενικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθυστέρησε όσον αφορά την παρουσίαση κατευθυντηρίων ε, γραμμών για την εφαρμογή της οδηγίας. Ο κύριος Καπούτο θα ήθελε να αναφερθεί σε διάφορα παραδείγματα του άρθρου 2 της οδηγίας ε, που περιορίζει το πεδίο εφαρμογής ε, και επιτρέπει τον αποκλεισμό κάποιων εγκαταστάσεων, αλλά ο αριθμός των εγκαταστάσεων που εξαιρούνται από τα κράτη-μέλη δείχνει ότι δεν ήταν σωστή η εφαρμογή. Ε, διάφορα κράτη-μέλη είπαν ότι δεν έχουν εγκαταστάσει κατηγορίας Α, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει εδώ εσφαλμένη ερμηνεία της οδηγίας. Γι' αυτό ο κύριος Καπούτο στηρίζει τον εισηγητή ε, που ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην καθυστερήσει κατά την παρουσίαση των κατευθυντηρίων γραμμών. Επίση, όσον αφορά το άρθρο 18 και τι σχετικέ εκθέσει από πλευρά ε, των κρατών μελών, ο κύριο Καπούτο λέει ότι από την ε, θέση σε εφαρμογή τη οδηγία οι ε, εκθέσεις που καλύπτουν τριετία έχουν υποβληθεί δύο φορές. Δεν είναι όμως συγκρίσιμα τα στοιχεία, διότι δεν υπάρχουν κατευθυντήρε γραμμέ σχετικά με την υποβολή των δεδομένων αν ανακοινωθούν τέτοιε κατευθυ... Ε, τέτοιες κατευθυντήρες γραμμές ε, θα έχουμε νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις ε, σχετικά με την υποβολή των στοιχείων. Επίσης, όσον αφορά τις επιθεωρήσεις, το άρθρο 32 προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει κατευθυντήρες γραμμές για τις επιθεωρήσεις, αλλά αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα και ως αποτέλεσμα οι διατάξεις για τις επιθεωρήσεις ερμηνεύονται διαφορετικά και εφαρμόζονται διαφορετικά στα κράτη-μέλη. Μια άλλη πτυχή που ο κύριος Καπούτο θεωρεί ότι αποτελεί προτεραιότητα σε διάφορα κρατημέλη είναι η εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για όλες τις εγκαταστάσεις κατηγορίας Α. Περίπου το 25% των εγκαταστάσεων δεν έχουν τέτοια σχέδια. Πράγμα που αποτελεί πρόβλημα και Τέλος, ε, όσον αφορά την κυκλική οικονομία, ε, το σχέδιο δράσης που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, προβλέπει νομοθετική αναθεώρηση της οδηγίας για τα εξορυκτικά απόβλητα. Και η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης των αποβλήτων και ο κύριος Καπούτο πιστεύει ότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει ε, συνολικό σχέδιο δράσης, διότι μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία καθώς και για το περιβάλλον. Και επιτρέψτε μου, κυρία Πρόεδρε, ε, ε, εγώ προσωπικά έχω κάποιες ερωτήσεις που θα ήθελα να θέσω στους εκπροσώπους ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει η διαδικασία επιπαραβάση κατά 18 κρατών μελών λόγω της αποτυχίας ή ελλειπούς εφαρμογή της οδηγίας στα στο εθνικό δίκαιο, αλλά θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας αναφέρει εναλλακτικά μέτρα που θα μπορούσε να λάβει στις περιπτώσεις αυτές. Και μια ερώτηση που έχει να κάνει με κάτι που ανέφερε και ο εισηγητής στις 5 ε, Μαΐου του 2010 στο ψηφίσμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο ε, ζήτησε νέα νομοθεσία, κάτι που απορρίφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρήθηκε ότι η ισχύουσα νομοθεσία αρκεί και το 2015 είχαμε άλλο ψήφισμα της, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, σχετικά με την καταστροφή της Ερυθράς ε, του 2010 και ε, εντόπισε τον τομέα αυτόν ως τομέα ιδιαίτερης ανησυχίας. Πιστεύουμε ότι και τα δύο αυτά παραδείγματα δείχνουν ότι ενώ έχουμε νέα οδηγία δεν μπόρεσαν να αποτραπούν καταστροφές και ότι δεν ολοκληρώθηκαν επαρκώς οι εργασίες στις περιπτώσεις αυτές. Επιπλέον, ανασχεδιασμός ε, του εργαλείου συλλογής ε, δεδομένων, μάλλον πέρα από το εργαλείο αυτό, τι άλλα σχέδια έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση αυτής της σημαντικής οδηγίας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάρκ Δεμεσμάκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ολλανδικά και ευχαριστώ τους εκπροσώπους ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και φυσικά και τον εισηγητή. Ήταν αρκετά εντελεχής ε, στην εισαγωγή του, γι' αυτό μπορώ να περιοριστώ σε λίγα λόγια, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Συμφωνώ με σχεδόν όλα όσα είπε. Συμφωνώ και με τις παρατηρήσεις του κυρίου Καπούτο που ακούσαμε από την κυρία Ντάλη. Δεν μπορεί να υπερβάλλει κανείς τη σημασία αυτή τη οδηγία. Τα εξορυκτικά και άλλα απόβλητα αποτελούν το 30% των συνολικών αποβλήτων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και συχνά μιλάμε για πολύ επικίνδυνα απόβλητα. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα την πορεία αυτών των αποβλήτων και για να έχουμε πιο κυκλική οικονομία. Ήδη τον Νοέμβριο πρότεινα τρει ε, προτεραιότητε όσον αφορά τη δική μα ομάδα. Βελτίωση τη ισχύουσα νομοθεσία, ε, βελτίωση τη υποβολή εκθέσεων και περισσότερη συνέπεια κατά την εφαρμογή από τι αρμόδιε αρχέ στα κράτη-μέλη. Οι προηγούμενοι ομιλητέ ήδη είπαν ότι οι μέσα από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αποτελούσαν βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Στο σχέδιο έκθεσης ο εισηγητής αναφέρει όλα τα θέματα αυτά και πιστεύω ότι η έκθεση αυτή αποτελεί πολύ καλή βάση για μας. Ακούσαμε και την αξιολόγηση σε της ε, εφαρμογής. Θα διαβάσω προσεκτικά τη μελέτη αυτή πιθανότατα να υποβάλω και σχετικέ τροπολογίε. Η έκθεση αυτή όμω, νομίζω ότι τονίζει τα σωστά σημεία. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Then um, another um, rapporteur, Madame Η κυρία Κονέτσνα, σκιώδης επίσης. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Επιτροπή γιατί μας ε, υπέβαλε πολλά στοιχεία τα οποία ε, έλειπαν. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή γιατί νομίζω ότι κατάφερε να εντάξει στην έκθεση όλα τα σημαντικά στοιχεία. Μια πολύ καλή βάση που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε όλοι και να συνεισφέρουμε έτσι ώστε να φτάσουμε στην ουσία. Αυτά τα απόβλητα, τα κατάλοιπα είναι ένα ουσιαστικό πρόβλημα είναι ε, πάρα πολλά αυτά τα κατάλοιπα τα οποία δεν μπορούμε να διαχειριστούμε σωστά. Η οδηγία ακριβώς θέλει να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα της αποθήκευσης ή εξάλληψης αυτών των καταλήπων. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολήθηκε με αυτό το θέμα εκ του σύνεγγης. Πολλά κράτη-μέλη μετέφεραν την ε, οδηγία πολύ σωστά, αλλά λιγότερο. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει η, ίση, η ίδια εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη, μια εναρμονισμένη προσέγγιση κατά τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία. Διαφορετικά θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον από τα κατάλοιπα αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία για να δούμε ποιες είναι οι ενδυνάμει απειλές. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα στοιχεία για να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων και οι επιπτώσεις του περιβάλλον όλες αυτές οι συνθήκες θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχει μια σειρά υποχρεώσεων για την αντιμετώπιση αυτών των καταλήπων. Θα πρέπει να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Η in situ έλεγχη είναι απαραίτητη για να δούμε πώς αποθηκεύονται τα κατάλοιπα αυτά. Θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή βάση λειτουργίας και εμπιστοσύνης. Ε, να μην μας ενδιαφέρει μόνο η αποκόμιση του κέρδους. Μιλάμε για επικίνδυνες ουσίες και οι αρμόδιες αρχές, οι ρυθμιστές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα με μεγάλη σοβαρότητα για να μην διατρέχουν κίνδυνο οι πολίτες. Διαφορετικά θα έχουμε να κάνουμε με μια ορολογιακή βόμβα την οποία δεν θα μπορέσουμε να απομονώσουμε. Δεν θα πρέπει να συγχαίουμε αυτά τα κατάλοιπα με κοινά κατάλοιπα. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα μέσα από τις μονάδες και τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης μεταξύ άλλων. Υπάρχει μια φιλανδική επιχείρηση η οποία εδώ και μερικά χρόνια ασχολήθηκε με τον έλεγχο παρομοίων περιπτώσεων και βλέπουμε ότι πολλές φορές το σύστημα μπορεί να αποτύχει. Γι' αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε και να συμφωνήσουμε για το ποια είναι η καλή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά την ασφάλειά μας. Και θα πρέπει να αποφύγουμε τους κινδύνους. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουν και την σωστή εντολή τα κράτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ε, συντάκτη και φυσικά θα συνεισφέρουμε ως οικειώδης όσο περισσότερο μπορούμε. Έκλεισε ο γύρος των ε, σχεδόν και η κυρία Πίρτερ έχει το λόγο. Ε, ζητώ συγγνώμη διότι ήταν, είχα μεγάλη δυσκολία και εγώ να φτάσω εδώ όπως και πολλοί άλλοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές και τον εισηγητή Προσβλέπω στην ε, ολοκλήρωση αυτής της έκθεσης και θα ήθελα να ε, μιλήσω για πτυχές ε, της εξόρυξης που αφορά το λεγόμενο seabed mining. Πολλά έχουν υποθεί για αυτόν τον τομέα ανά τον κόσμο. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι πόροι που έχουν επενδυθεί, αλλά έχει, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η εξόρυξη στη θάλασσα δεν είναι τόσο δαπανηρή. Και εδώ, ε, από όσο γνωρίζω, στη Βόρεια Θάλασσα υπάρχουν πολλά κοιτάσματα άνθρακα ιδιαίτερα και πολλές φορές είναι δύσκολο να μεταφερθούν αυτά τα μέσα σε άλλα μέρη του κόσμου, διότι ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλές φορές αυτή η εξόριξη είναι πολύ πιο εύκολη στην επιφάνεια της θάλασσας. Επίσης, όταν ε, ασχολήθηκα με την τοπική αυτοδιοίκηση, είχαμε πολλές ε, χωματερές όπου ε, ποντίζονταν υλικά τα οποία δεν επιτρέπεται πλέον να ποντίζονται. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Θα δείτε ότι στο Johannesburg ε, γύρω από την πόλη υπήρχαν ε, χωματερές και είχαμε να κάνουμε εκεί με κατάλοιπα χρυσού τα οποία βρίσκονταν στην περιφέρεια του Johannesburg. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι χωματερές που έχουμε ε, στην Ευρώπη θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αλλιώς μέσα στα πλαίσια αυτών των καταλήπων που δημιουργούνται και αποθηκεύονται. Και εδώ μιλάμε για εφαρμογή της νομοθεσίας. Αυτό είναι το θέμα ουσίας γιατί η νομοθεσία είναι πολύ καλή, νομοθετούμε πολύ καλά, αλλά είναι πολύ δύσκολο να επιθεωρήσουμε in situ την εφαρμογή της νομοθεσίας. Και αυτό αφορά και τη δραστηριότητα της Κομισιόν, δηλαδή πολλές φορές γίνεται επίβλεψη, αλλά μετά, τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια ε, μετά και δυστυχώς βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα είναι ολέθρια μετά από πέντε χρόνια. Και ιδιαίτερα σε μικρές ομάδες βλέπουμε ότι πολλές φορές υπάρχουν σημαντικές ε, επώδυνες επιβλαβείς επιπτώσεις, όπως ακούσαμε και από πολλά κράτη-μέλη, τα οποία δυστυχώς δυστυχώς ε, δεν έχουν ε, εφαρμόσει αυτές τις ε, οδηγίες. Λυπάμαι που ο Σκιώδης δεν είναι παρόν, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να φτάσει μέχρι εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα τώρα οι εμπειρογνώμονες κάτι να προσθέσουν, αν έχουν κάτι να προσθέσουν σε όλα όσα υπόθηκαν. Έχετε το λόγο. Δεν είμαι βέβαιος ότι κατάλαβα τι ερωτήσεις σας γιατί σε μεγάλο βαθμό πρώτα περί σχολείων, μιλήσατε για το seabed mining. Εγώ δεν μπορώ να σας πω κάτι. Τουλάχιστον ε, μπορώ να πω κάποια πράγματα, δεν είμαι αυθεντία στα θέματα της εξόριξης ε, του βυθού. Όμως υπάρχουν και κάποια άλλα στήματα. Και υπάρχουν και διεθνή εργαλεία και κανονιστικά μέσα μάπολη, κάτι τέτοιο και πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη, αλλά επαναλαμβάνω δεν είμαι εμπειρογνώμη, δεν είμαι η για αυτά τα θέματα. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε για τους δευτερογενείς πόρους ή ε, πρώτες ύλες, ε, οι χωματερές ή τέλο πάντων απόβλητα ορυχείων εν γέννη. Αυτό που χρειάζεται κατά την άποψή μου είναι μια πιο συστημική θεώρηση για το πώς παρέχουμε πρώτες ύλες στις κοινωνίες μας. Αν, ε, για παράδειγμα, δείτε τι έγινε και τι γίνεται μάλλον σήμερα στην έρευνα, θα δείτε ότι ακριβώς αυτό επιδιώκουμε. Να δούμε πού παίρνουμε μεταλλεύματα, πρώτες ύλες από ορυχεία εδώ ή ε, εξωχώρια Επίσης υπάρχουν δευτερογενείς πηγές, οματερές και άλλα σημαία αναπόθεσης βλήτου. Συμμετέχω και εγώ λοιπόν σε αυτές τις προσπάθειες, σε αυτή την έρευνα και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να το συνδυάσουμε αυτήν την προσωπική μου άποψη με την οδηγία για τα απόβλητα ορυχείων, διότι κατά πάσα πιθανότητα πολύ σύντομα το ξέρετε και πολύ καλά, θα φτάσουμε σε μια ε, φάση που δεν θα λέμε τα απόβλητα απόβλητα. Απλά είναι ύλες οι οποίες κάπου έχουν αποτεθεί προσωρινώς και η χρήση για αυτά τα υλικά θα, ε, θα υπάρξει μάλλον κάποια χρήση για αυτά τα υλικά κάποια στιγμή. Τώρα σε τις μονάδες ε, τα λοιπά. Υπάρχουν κάποια προβλήματα με την ορολογία. Legacy, site λοιπά. Εγώ είμαι Γερμανός, αλλά μου ξέρω και για την Αγγλία. Υπάρχουν κάποιες εγκαταστάσεις ε, που χρονολογούνται εδώ και αιώνες. Ήταν κάποια μεταλλορυχία, κατά το παρελθόν περιλαμβάνουν τώρα μεταλλεύματα που τα γνώριζα μεν ο κόσμος, αλλά δεν μπορούσε ίσως να τα αναγνωρίσει και μπορεί να μην ξέρουμε αν καλύπτεται κάποιο συγκεκριμένο μετάλλευμα από την οδηγία ή όχι. Και σε παλαιότερα τέτοια ορχεία, πού βάζουμε το όριο. Είναι ιστορική εγκατάσταση, όχι. Ε, και πιστεύω ότι όταν χαρτογραφηθούν ε, και οι πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές πρώτων υλών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει αυτά να μπουν ίσως στην ίδια θέση. Και θα πρέπει να ποια είναι τα μεταλλεύματα ε, δημόσιο ενδιαφέροντος και πώς μπορεί να γίνει εξόριξη και ίσως λυθούν και κάποια προβλήματα ταυτόχρονα που αφορούν τα πόβλητα. Η χαρτογράφηση όμως είναι ένα πρόβλημα και έχουμε και κάτι ακόμη. Το πρόβλημα της αδειοδότησης για εξόριξη Αναφερθήκατε στις χωματερές που είναι κοντά σε αστικές περιοχές περισσότερες ε, περιπτώσεις. Πώς θα δοθεί λοιπόν δημόσια συγκατάθεση παρότι αυτό για εξόριξη, παρότι μπορεί τα ωφέλη για την κοινωνία να είναι ξεκάθαρα. Θα είναι δύσκολο. Είναι πολύ διάστατο λοιπόν το πρόβλημα. Γιατί έχει τεχνικά ζητήματα, ρυθμιστικά και προβλήματα δημόσιας αποδοχής. Σας ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο του στον κύριο Λάγκετορφ, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη που καθυστερήσαμε, δεν γνωρίζαμε ότι εξετάσατε νωρίτερα το θέμα αυτό. Ελπίζω όμως να ενημέρωσαν επαρκώς οι συναδελφοί μου, ώστε να μπορέσω να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις. Κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με την έκθεση και το ψήφισμα. Πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμα για τη δουλειά μας και πολλές από τις συστάσεις στο σχέδιο ψηφίσματος αναφέρονται σε δουλειά που ήδη κάνει η Επιτροπή. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ευθυγραμμίζεται πολύ καλά η δουλειά μας με τις συστάσεις. Όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, υπήρξαν κάποια προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν ε, ακόμα κάποια προβλήματα, πιστεύουμε όμως ότι θα λυθούν σύντομα. Έχουμε εντοπίσει τα προβλήματα που υπάρχουν και τα κράτη-μέλη μας έχουν υποβάλει νέα κείμενα σχετικά με την εφαρμογή. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτό το θέμα βρίσκεται υπό έλεγχο. Όσον αφορά την ευρύτερη εφαρμογή της οδηγίας, πέρα από την ε, εφαρμογή και τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, ε, υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης δικαστικής δράσης, κάτι που έχει γίνει κατά κάποιων κρατών μελών. Νομίζω ότι αυτό απαντάει και σε κάποια από τις ερωτήσεις που τέθηκε. πέρα από τις ε, δικαστικές ε, ενέργειες. Συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές, ε, να δούμε τι μαθήματα μπορούμε να εξάγουμε. Θα πραγματοποιηθεί σημαντικό εργαστήριο τον Μάρτιο του 2017, φέτος τον Μάρτιο, το οποίο θα μπορέσει να παρακολουθήσει όποιος ενδιαφέρεται και θα ακολουθήσει μια μελέτη στο δεύτερο εξάμεινο του χρόνου που θα εντοπίζει τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τα αποβλητά ορυχείων. Επίσης, ε, θα εκπονήσουμε κατευθυντήρες γραμμές σχετικά με τις βασικές έννοιες της οδηγίας ε, για να διασφαλίσουμε την ε, πιο συνεπή εφαρμογή. Αυτές λοιπόν είναι οι πτυχές της δουλειά μας, ε, συμμόρφωση, προώθηση και κατευθυντήρες γραμμές. Στο σχέδιο ψηφίσματος, όπως άλλωστε αναφέρεται, εργαζόμαστε πάνω στις κατευθυντήρες γραμμές ε, για τις καλύτερες επιθεωρήσεις. Θέλουμε τις ε, περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις να τις συμπληρώσουμε με κατευθυντήριες ε, γραμμές ειδικά για την ε, εξορυκτική βιομηχανία ε, και ελπίζουμε να εκπονηθούν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές του χρόνου το αργότερο. Επίσης, στο ψήφισμα αναφέρεται η υποβολή εκθέσεων. Θα θυμάστε ότι το Νοέμβριο Σας υποβάλαμε έκθεση σχετικά με την ε, έκθεση εφαρμογής της οδηγίας ε, που καλύπτει την εφαρμογή τα τελευταία χρόνια. Ε, δεχόμαστε ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων, τις οποίες θέλουμε να καλύψουμε. Αυτό αποτελεί μέρος ε, του fitness check που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας συνδέεται στενά και με άλλες οδηγίες, ε, την ε, οδηγία για τις εκπομπές για παράδειγμα. Εξετάζουμε πώς μπορεί να απλοποιηθεί η διαδικασία υποβολής εκθέσεων, μειώσουμε το διοικητικό άχθος όπου μπορεί να γίνει αυτό και αυτή είναι μια συνεχιζόμενη προσπάθεια. Στο μεταξύ, όπως ε, σας είπα, Έχουμε την μελέτη σχετικά με την ε, συμμόρφωση και την ε, μελέτη που πραγματοποιούμε αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά την απαγόρευση κυανιδίων, Θα σας παραπέμψω στην απάντηση που έχει δώσει επανειλημμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάγκη για τέτοια απαγόρευση, δεδομένου ότι η οδηγία παρέχει επαρκή εχέγγυα για την ασφαλή χρήση κυανιδίων, συμπεριλαμβανομένων πολύ αυστηρών οριακών τιμών. Σας παραπέμπω σε απαντήσεις που σας έχουμε δώσει και το 2012 και το 2015 και πολύ πρόσφατα σε απάντηση ε, αιτήματος πάνω στο θέμα αυτό αναφοράς ε, που θα συζητηθεί μάλιστα αύριο στην Επιτροπή Αναφορών. Ερωτήθηκε αν υπάρχουν πιο αποτελεσματικοί τρόποι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα κατά την εφαρμογή. Έχουμε λοιπόν τις ε, παράλληλες διαδικασίες, συμμόρφωση προώθηση της συμμόρφωσης και δικαστική δράση όπου αυτό είναι απαραίτητο. Βέβαια, η... αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει τη μόνη αντίδραση. Όσον αφορά τις χωματερές, ε, την οδηγία για την εξορυκτική βιομηχανία, είναι θέματα που καλύπτουμε και στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία. Συγκεκριμένες δράσεις ε, στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία αναφέρεται στην οδηγία για τα απόβλητα ορυχείων. Επίσης, έχουμε συμπληρωματικές εργασίες που έχουν να κάνουν με την ε, βελτίωση της νομοθεσίας ε, και του κανονιστικού πλαισίου. Αναφερόμαστε και, στα και στις δευτερογενείς πρώτες ύλες ε, που προκύπτουν από τα απόβλητα ορυχείων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα έχουμε αυτά αποτελέσματα μέσα στο επόμενο έτος. Ελπίζω ότι έτσι απάντησα σε κάποιες από τις ερωτήσεις. Αν υπάρχουν και άλλες, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή για να κλείσει τη συζήτηση. Δεν είναι απαραίτητο. Ωραία. Κύριε Καπούτο, όχι. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση αυτή. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 14η Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Έτσι ολοκληρώνονται οι σημερινές μας εργασίες. Θα σας δω όλους αύριο το πρωί στις 9. Σας ευχαριστώ πολύ.